Καλημέρα σας, να ξεκινήσουμε. Bene, buongiorno a tutti. Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής, τη Γραμματεία, τους βοηθούς. Πιστεύω ότι χθες δείξαμε, όπως να γίνει και σήμερα με την έκθεση του κυρίου Λαβία, δείξαμε ότι η Επιτροπή μας ε, κατόρθωσε να ψηφίσει και ξεκάθαρα να παρουσιάσει τις ιδέες της για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τους κοιόδης και τη γραμματεία. Και φαντάζομαι τώρα ότι ο Τζεβάνι θα θέλει να πάρει το λόγο πριν να ξεκινήσουμε με το τελευταίο από τους τελευταίους νομοθετικούς φάκελους για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Παρακαλώ, κύριε Σλαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω ένθερμα τους Σκιώδης, ε, τους ε, υπαλλήλου των πολιτικών ομάδων και τη γραμματεία που μα συνόδευσαν σε όλη αυτή τη διαδρομή τροποποιήσεων της πρότασης της Κομισιόν για τον οριζόντιο κανονισμό. Ήταν ε, μακρά η εργασία και πολύπλοκη, καθώς είναι ιδιαίτερα τεχνικός ο κανονισμός αυτός και σήμερα με την ψηφοφορία ολοκληρώνεται αυτή η εργασία. Και φυσικά απευθύνω τις ειλικρινές ευχαριστήσεις μου σε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου, από τους βοηθούς μέχρι τους υπαλλήλους ε, και τα, τους υπαλλήλους γραμματείας, αλλά και σε όλες τις άλλες ομάδες, γιατί θεσπίστηκε μία πραγματικά ειλικρινή σχέση συνεργασίας ε, που κατόπιν ε, αντικατοπτρίστηκε και στι συμβαστικέ τροπολογίες τι οποίες συμφωνήσαμε και ελπίζουμε σήμερα να μπορούν να ψηφιστούν, να υπερψηφιστούν από όλε τι πολιτικές ομάδε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε του ίδιου κανόνε με χτε. θα ψηφίσουμε όλους ε, τους συμβασμού με ηλεκτρονική ψηφοφορία και με ένα τασιχυρό όλα τα υπόλοιπα, Όλε τι υπόλοιπε τροπολογίε. Είμαστε έτοιμοι. να ξεκινήσουμε με το άκρο 7 του εισηγητή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία budget 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές, Απορρίπτεται θα έλεγα. 176 έκουτ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος μάλιστα. Για το 176 άρχεται η ψηφοφορία. το όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Υπολογία 11 το συγκητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 178 νταντέν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 180 Ντόρφμαν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 γκίρλινγκ υπέρ κατά αποχές έλεγχος με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 183 Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 186 άντρου τραμπέλα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 του συγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολμέιρ 188 υπέρ, κατά. Μάλλον πρέπει να ελέγξουμε την 188. Εγκρίνεται. Για μία ψήφα. Κόντα 6. Περ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 194 του συγητή. Υπέρ. Κατά αποχές. εγκρίνεται. 191 δες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κόντ 7 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Κόντ 7 Ψήσατε όλοι. Εγκρίνεται. Κόντο 8 πέρ Κατά. Εποχές. Και εδώ έλεγχος για το 8. Εγκρίνεται θα έλεγα. Ναι. 195 ρούμπι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 197 Μάιερ υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για το συνδεσμό 1 η ψηφοφορία Συμβασμός Πετμόν 1. Βλέπω εδώ τους πρασίνους, θα έλεγα, μάλλον βλέπω πράσινα τα λαμπάκια, θα έλεγα εγκρίνεται. Μάλιστα, πάλι με ηλεκτρονική ψηφοφορία, στο συμβασμό υπάρχουν δύο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Κάνουμε ένα άλμα και πάμε στην τροπολογία 26 του συγητή υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.72 ντύσεκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά για το συμβασμό 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα να περάσουμε στην 78. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο. 79 φαϊμών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 280 δανέλης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 Μάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 283 καρόνα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 285 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 31 του εισηγητή υπέρ κατά εποχές έλεγχος για την 31 θα έλεγα πόσο εγκρίνεται, αλλά για να δούμε μάλιστα κρίνεται 2.87 εκούτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα με ηλεκτρονική ψηφορία Άρχεται η ψηφορία για το συμβασμό 4. Ψήφιζε όλοι. Εγκρίνεται. Τώρα, ένα τεσσεχειρός 2,89 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 33, του συγητή υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. Τώρα 35 του συγητή υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 291 δες υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 36 του συγητή υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 38. Πάλι το συγγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρακόσια τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 307 Δίας Δαμέρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Έναν έλεγχο να κάνουμε για το 307. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα έλεγα ότι απορρίπτεται λίτερο πρόεδρος. Πέρας. Ναι. Απορρίπτεται. 310 ντούσεκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 309 γκίρλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 313 νταντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 314 γκουτιέρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 του εισηγείται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 319 Νταντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 320 Καρόνα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 327 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτω. Θέλετε έλεγχο για το 327. Μάλιστα. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν υπήρχαν αμφιβολίες. Απορρίπτεται. Τώρα, μένοντα ηχηρό, 334 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 336 τριάντα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για το 336. Μάλιστα, εγκρίνεται. 3.38, με ένα τασχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα πως εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για την 3.38, παρακαλώ. Είμαστε πολύ κοντά, μία-δύο ψήφι διαφορά από ό,τι φαίνεται. Ψήφισατε όλοι. Ναι, απορρίπτεται. Λοιπόν, 3,47 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για το 3,47. Εγώ θα έλεγα πως απορρίπτεται. Ε. Ψηφίσατε όλοι. 347. Απορρίπτεται. Ευραίος. 350. Λάιον. Περ. Μετά ισχυρός. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το έχουμε βρει πλειοψηφία υπέρ. 349. τα ισχυρός υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 του συγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 353 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο για την τροπολογία 353. Θα έλεγχο που εγκρίνεται. Απορρίπτεται για μία ψήφο. 352 Χολμάιερ. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 354 Σάρμπου. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 του σιγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 20 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Υπάρχουν αμφιβολίες έλεγχος για τη Ρέτζι 20 παρακαλώ. Απορρίπτεται. Τα έλεγα, αλλά σε ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Μάλιστα. Όντως. 3.56 Ρούμπιξ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 357 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα εγκρίνεται ελέγχουμε για τη 3.57 άρχεται ψηφορία ψήφισατε όλοι απορρίπτεται Πάμε με ναι, τεσχυρό πάλι στην κόντ 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται θα έλεγα. Κόντ 15. Υπέρ. Κατά. Και εδώ εγκρίνεται. 16 κόντ υπέρ κατά εγκρίνεται 47 του εισηγητή υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 365 λάϊον υπέρ κατά εγκρίνεται 48 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 372 Λάιον υπέρ κατά Αποχές. εγκρίνεται 374 υπέρ Κατά. εποχές εγκρίνεται. Κοντ 19. Υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. 376 υπέρ. Κατά. εποχές εγκρίνεται. Κόν 21. Υπέρ. Κατά. Εποχέ, εγκρίνεται. 54 του συγγητή υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται. 379 γκίρλινγκ υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται. Τώρα, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, συμβιβασμό 5, άρχεται ψηφοφορία. Τι. Ψηφίσατε όλοι. Έγκρινεται. Πάμε στην 391. Δυνατά στους υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 392 του ΖΕΚ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 407 υπέρ. Όχι, συγγνώμη λέει ο μισό λεπτό. Πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την 401 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 407 Holmeyer, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για την 57 ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 57 πέρας εγκρίνεται. Κόντι 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 414 ντούσεκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κόντι 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 416 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 του συγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 417 υπέρ κατά Εδώ πρέπει να γίνει έλεγχος για την 417 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πρέπει να είναι θετικό το αποτέλεσμα, αλλά ας δούμε. Ψηφίσατε Μάλιστα, εγκρίνεται. 59 το εισηγητή. Διανατάσεις ισχυρός υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία στη συμβαστική τροπολογία 6. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Συγχαρητήρια. Συμβαστική 6 έτυχε της πλήρους υποστήριξης. Πάμε στη συμβιβαστική 8. Συνάδελφοι, ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική 8. Ψηφίσατε όλοι. Και εδώ έχουμε μεγάλη πλειοψηφία. Υπέρ. Τρο... χειρός στην 73 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 450 Μάιερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 του εισηγητου 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 9. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Δυνατές 458 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 460 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 461 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 462. 462 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 462 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Εγώ θα έλεγα ότι με μικρή διαφορά εγκρίνεται. Ναι, εγκρίνεται. 463 αριαντές του χειρός υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 465 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 467 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 468 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 469 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 470 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 471 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 473 Σίμψον υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, συνάδελφοι, για τη συμβαστική 10. Ξεκινάει ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δυνατάς ισχυρός. Τροπολογία 479 Αλετζνέκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Και εδώ με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ως συνήθως ξεκινάει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. εγκρίνεται. Κάνουμε ένα μικρό άλμα και πάμε στην 84. Δυνατάσως χειρό. Τροπολογία 84 του συγητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 510 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 511 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 512 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 513 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 514 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, διαλεκτρονικής ψηφοφορίας, την συμβαστική 13, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Διανατάσεις της χειρός 520 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Andiamo Πάμε στην 527 του συγκριτή υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 528 άρκιν υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να κάνουμε έλεγχο στα γρήγορα. 528 Χάρκιν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 529 Μάιερ υπέρ, κατά, κατά, αποχές, πρέπει να κάνουμε έλεγχο. 529 Μάιερ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. 530 δυνατά στο χειρός. 530 του συγκητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 532 Άρκιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 533 δυνατά στους χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 536 σάρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 537 λάιον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 540 για υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 543 γκέρλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 545 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 546 έκχουτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 547 Ιάρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 548 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 549 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 550 έκχουτ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 553 γκέρλινγκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 559 μαγκίνες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 562 λάιον υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 558 δελάνς υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 560 ντούζεκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 561 φαϊμόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στη Ρέτζη 27. Ρέτζη 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 564 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 565 Lion υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 566 Νικουλέσκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 88 του συγητού υπέρ, κατά, αποχές, απο, εγκρίνεται, συγγνώμη. Όχι, έλεγχος. 88 του εισηγητού, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Για να 89 του συγητού. 89 υπέρ. Κατά. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο. 89. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 587 διανατάς χειρός υπέρ. Α, πάμε στη συμβαστική 14 ηλεκτρονική ψηφοφορία που άρχεται για τη συμβαστική 14. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, εγκρίνεται. 593, δυνατά στους χειρός, 593 ήταν υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 594 Νικουλέσκου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωται. 595 Ταντέν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτωται. 597 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90 του συγητού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 609 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 611 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 601 ροντ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 του συγητού υπέρ, κατά, αποχές, θα έλεγα ότι εγκρίνεται. 602 έκχουτ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 603 ο Λετζινζάκ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 606 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 28, δυνατές χειρός υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 604 Simpson υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 607 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 608 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 610 χάρκιν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 612 μαέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 94 του συγγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 617 ο Νίτσακ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική 15. Ψηφίσατε όλοι. Η συμβαστική 15 εγκρίνεται. Ένα αλματάκι Πάμε στην 640 δυνατά του υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να κάνουμε έλεγχο. Είδα πολλά χέρια. Παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 640 εράνς. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται. Πάμε στην 639. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέτζι 30. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 646 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συμβαστική 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Διανατάσσεως χειρός 647 έραντζ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 649 γιάρ υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Για την 649 ηλεκτρονικός έλεγχος. 649 γιάρ. Νομίζω ότι πρέπει να εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφόριας, εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική για τη συμβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ομόφωνα εγκρίνεται. Πολύ καλά. Τροπολογία 655 Μάιερ. Ανατάσσεται χειρό υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 97 του συγητού υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική για τη συμβαστική 18. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 661. 661. Δυνατά σειρό υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 662 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύε 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 676 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 677 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 678 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στη διαφάνεια. Ξεκινάμε με την 803 δες για Κατά. Έλεγχος. Για την 803 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα την τροπολογία 788, 788 του συγκριτού υπέρ, κατά αποχές. Ας κάνουμε έναν έλεγχο και εδώ σας παρακαλώ, γιατί την 788 ηλεκτρονικός έλεγχος. 788, πέρας. Εγκρίνεται. 813 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 815 Ανδρέο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 816 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός για την 816 Ανδρέου σας παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 679 του συγκητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 681 Μάιερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 684 Νικολέσκου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 685 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 686 υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον εγκρίνεται. 687 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 688 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 689 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 690 Reimers υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 691 Έκχουτ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 692 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 693 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 694 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 695 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 696 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 697 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 698 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 699 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 700 Ράιμερς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 701 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 702 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 703 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 704 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 705 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 706 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 707 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας γίνει έλεγχος για την 707 εράν σας παρακαλώ πολύ. Ψηφίσατε όλοι. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. 708 κουτιέρες υπέρ 708 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 710 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 714 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 715 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Συγγνώμη λοιπόν. 715 δαντέν ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίνεται λοιπόν η 715 δαντέν. 716. Α όχι. Πάμε στην 717 έκχου τυπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 718 υπέρ κατά έλεγχος για την 718 σας παρακαλώ 718 ντες έλεγχος πέρας εγκρίνεται 721 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλετε έλεγχο στην 721 ζητήθηκε ηλεκτρονικός έλεγχος για την 721 δες άρχεται η ψηφοφορία εγκρίνεται Πάμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία στη συμβιβαστική 19. Συμβιβαστική 19, ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. 726 δες πάμε τώρα. 726 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 700... 700 Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική 20. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, συμβιβαστική 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Διανατάσσου της χειρός 745 έγχουτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία της συμβαστική 22. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Διανατάσσω της χειρός. 752. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 753. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 775 Davis υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 754 Danten υπέρ, κατά, κατά, αποχές, μάλλον εγκρίνεται. Έλεγχο σας παρακαλώ. Έλεγχος για την 754. Εγκρίνεται λοιπόν. Η, η 754 εγκρίνεται. 755. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 756 Δες, υπέρ. Υπέρ. Τις 756 κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 756. Θα γίνει έλεγχος ηλεκτρονικός σας παρακαλώ για την 756. Εγκρίνεται. 758 δυνατές σειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 759 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ξεκάθαρο τι έγινε με την 759 DES, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 759. Εγκρίνεται. «760 τώρα, δυνατά στους γυρός υπέρ». «Κατά». «Αποχές». Μάλλον εγκρίνεται. 761 υπέρ. Όχι, την αφήνουμε. 762. 762 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ θα έλεγα ότι εγκρίνεται. 765 έραν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 766 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 768 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύε 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 Κάντεμπαχ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105 Ολμάιερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1. Τροπολογία 1 του συγητού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 2 Έλεγχος υπολογισμού 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εισηγητού 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107 άρκιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 γκέρλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109, α, συγγνώμη, 111 All Reaper κατά αποχές εγκρίνεται. Να κάνουμε ηλεκτρονικό ελέγχο για την 111. Εγκρίνεται λοιπόν. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Πάμε διανατάσσω στις χειρός στη Ρέτζι 3. Η Ρέτζι 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117 έκθοτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη Ρέτζι 5 υπέρ. Ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 Γκέρλινγκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 Άρκιν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 Λάιον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 όλμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δυνατάς χειρός, Τροπολογία 136. Βαϊτσεκόφσκι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε δυνατά χειρός στην 142. Γκέρλινγκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Υπέρ, για τη Ρέτζη 10. Συγγνώμη, υπέρ, εγκρίνεται. Η Ρέτζη 10 εγκρίνεται. 143 Λάιον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 του συγητού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Infatti. Per dubbio, meglio votare. 152. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για την Dorfman 152, ηλεκτρονικός έλεγχος. 152 λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε με μία ψήφο. Διαφορά. Μπράβο, Dortmund 152. Ψηφίζουμε την 157 γιάρ, δυνατά στους γυρός, 157 υπερ, κατά. Ένας έλεγχος και εδώ θα έλεγα, παρακαλώ συνάδελφοι. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 157 γιάρ. Ψηφίσατε όλοι. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Ας ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Πάμε στη Ρέτζι 11. Δυνατά σχηρό υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 164 χάρκιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167 Ολενίτσακ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168 Λάιον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αμφιβολίες για την 168 ηλεκτρονικός έλεγχος σας παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ρέτζι 12, διανατάσεις χειρός υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 171 171 εγώ θέλω ότι απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος όχι εγκρίνεται 172 Eichhut υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 790 Ανδρέου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 780 του σιγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελευταία σελίδα 781 του συγκητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 798 Ανδρέου, διατάσσει χειρό υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 799 για υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 800 Ανδρέου υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη λέει ο πρόεδρο. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 801 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση αυτή με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για να ξεκινήσουν οι διοργανικές διπλωματές. Ψηφίσατε όλοι. Σας ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία όσον αφορά τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και να χειροκροτήσουμε τον εισηγητή Τζοβάνι Λαβία. Συγχαρητήρια σε εκείνον, σε όλους τους εισηγητές. Στον Γιώργο Παπαστάμκο που έδωσε τη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό και σε όλους τους συναδέλφους σας ευχαριστώ για την έξοχη δουλειά. Συνάδελφοι, προσοχή παρακαλώ. Έχουμε πάνω από μία ώρα διάλειμμα, αλλά θα πρέπει να τα ξαναπούμε εδώ στις 11.30, διότι έρχεται ο κ. Σοφοκλής Αλετράρης, ο Υπουργός Γεωργίας της Κύπρου, που ε, είναι η επερχόμενη Προεδρία, που θα κάνει την αποτίμηση της εξερχόμενης Προεδρίας Έχουμε μία ώρα και 15 λεπτά για διάλειμμα. Παρακαλώ να έρθετε εδώ στις 11.30. Σας ευχαριστώ όλους. Siamo. Bene. Να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε όλοι. Και έχω την ικανοποίηση να καλωσορίσω για μια ακόμη φορά τον φίλο, τον κύριο Υπουργό Γεωργίας ε, της Κύπρου, τον κύριο Σοφοκλή Λετράρη τέλεση πρόεδρος του Συμβουλίου Γεωργίας, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωργίας ε, και σήμερα θα μας προσθέσει τα αποτελέσματα της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας. Ήταν ε, σημαντικό το έργο που υλοποιήσαμε κατά το εξάμεινο της Κυπριακή Προεδρίας. Ε, είχαμε πολλές συζητήσεις, επίσημες και άτυπες, άτυπους τριμερείς διαλόγους που νομίζω ότι βοήθησαν πάρα πολύ στην αμοιβαία ε, συνεννόηση του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου και μας βοήθησαν και να καταλήξουμε και στις αποφάσεις μας. Και μάλιστα ψηφίσαμε χθες και σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας τους τέσσερις νομοθετικούς φακέλους που αφορούν τη μεταρρυθμίση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα καταφέρουμε και σημειώνοντας και ευρεία πλειοψηφία και ξεπεράσαμε το 70% των ψήφων σε όλους τους φακέλους. Ε, είμαι λοιπόν πολύ ικανοποιημένο ε, και εγώ νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να μπορέσουν να σημειώσουν πρόοδο με το έργο της ε, Κυπριακής Προεδρίας, να συνεχιστεί αυτό το έργο υπό την Προεδρία της Ιρλανδίας, έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σου εδώ και τη διαθεσιμότητά σου και σε ευχαριστώ που σε τόσες πολλές περιπτώσεις ε, μας έδειξες ε, πόση σημασία δίνει η Κυπριακή Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Με μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν θα σου δώσω το λόγο και κατόπιν της παρέμβασής σου θα ζητήσω από τους επικεφαλείς ε, των ομάδων, από τους συντονιστές και οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο να πάρει το λόγο αν το επιθυμεί. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση που βρίσκομαι σήμερα και πάλι μαζί σας για να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της γεωργίας και ειδικότερα για την πρόοδο που επετεύθηκε στην εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής για μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Στις 10 Ιουλίου του περασμένου χρόνου, όταν είχαμε την πρώτη μας συνάντηση, σας διαβεβαίωσα ότι η Κυπριακή Προεδρία προσέβλεπε σε παραγωγική συνεργασία με θετικό πνεύμα και καλή θέληση ανάμεσα στα δύο θεσμικά μας όργανα, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για πρόθεση των κοινών στόχων στον τομέα της ευθύνης μας. Θέλω σήμερα να σας ευχαριστήσω για τη στενή αυτή συνεργασία η οποία υλοποιήθηκε με τις τρεις παρουσίες και ομιλίες μου ενώπιον της Επιτροπής σας και με τους τρεις ούτω καλούμενους Anticipatory Trialogues που πραγματοποίησαμε στις 9 Σεπτεμβρίου, στις 11 Οκτωβρίου και στις 6 Νοεμβρίου στην παρουσία του Επιτρόπου Σιόλου και με τις πολλές άλλες ανεπίσημες συναντήσεις και επαφές που είχαμε σε άλλα επίπεδα. Σημειώνω ειδικότερα ότι ο Πρόεδρος της ειδική Επιτροπής Γεωργίας, ενεργώντας εκ μέρους του Συμβουλίου, πραγματοποίησε με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής εννέα συνολικά θεσμοθετημένους τριλόγους με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. Μόλις στις 4 Ιουλίου 2012, τέσσερις μόνο μέρες μετά την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο, καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία σε σχέση με τον κανονισμό για τη στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές. Στο μεταξύ, τόσο ο κανονισμός αυτός όσο και ο άλλος μεταβατικός κανονισμός που ρυθμίζει τις άμεσες πληρωμές για το 2013 έχουν ψηφιστεί από τα δύο μας σώματα και έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Το ίδιο έγινε και με τον κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για τον οποίο έχει επιτευχθεί συμβιβασμός επιδανικής προεδρίας. Εξάλλου, το πολύ θετικό πνεύμα που επικράτησε κατά τους τέσσερα συνολικά τριλόγους που είχαμε για τους κανονισμούς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε τα γνωστά προβλήματα περιλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με την ευθυγράμμιση με την συνθήκη της Λισαβόνας και να επιτύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2012. Άξια αμνίας είναι επίσης και η συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο σε σχέση με τους κανονισμούς για τους αρωματισμένους ίνους όπου πετύχαμε αποφασιστική πρόοδο μετά από τρεις γύρους τριλόγου και καθώς και για τον κανονισμό για τα λογιστικά στοιχεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπου κάναμε μια καλή αρχή. Το ίδιο ισχύει και για την πρόταση κανονισμού για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, όπου επιτεύθηκε σημαντική πρόοδος για πολλές από τις προταθήσεις τροπολογίες και δημιουργήθηκαν καλές προοπτικές για επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Η Κυπριακή Προεδρία ετοίμασε επίσης συμβιβαστική πρόταση κειμένου για την ηλεκτρονική αναγνώριση βοηδών και την απάλληψη των προνοιών για την εθελούσια σήμανση με βάση την οποία δόθηκε εντολή στην Ιρλανδική Προεδρία στις 11 Ιανουαρίου 2013 για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο. Στον χτινιατρικό τομέα η Κυπριακή Προεδρία είχε επίσης την ευκαιρία να διοργανώσει δύο σημαντικά διεθνή συνέδρια για επίκαιρα θέματα. Το πρώτο αφορούσε την εισαγωγή και διατήρηση των εξωτικών ζώων στην Ευρώπη και το δεύτερο την προστασία των ζώων στα σφαγεία κατά τη στιγμή της σφαγής. Ολοκληρώνω την αναφορά μου στην πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων και με την Επιτροπή επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας επετεύθηκε σε πρώτη ανάγνωση η ψήφιση των δύο αποφάσεων που αφορούν τους πόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό και δεν τέθηκε σε κίνδυνο η εισαγωγή των ειδών αυτών από τρίτες χώρες μετά από την 1η Πρώτου 2013. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου τώρα να επικεντρωθώ στα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Μιλούμε για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση σε εύρος και σε βάθος, για την οποία όλοι είχαμε εξ αρχής τη συνέστηση ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα πλαίσια των συζητήσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Ως Προεδρία είχαμε ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι υπήρχε ανάγκη να επιτύχουμε χειροπιαστή πρόοδο το ταχύτερο δυνατόν γιατί τα χρονικά περιθώρια που μας είχαν απομείνει προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη συμφωνίας και η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ από 1η 1η-1η 2014 ήταν ήδη πάρα πολύ στενά. Κατά συνέπεια, θέσαμε εξ αρχής ως στόχο την επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο προκειμένου το Συμβούλιο να είναι σε θέση να αρχίσει επίσημες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την αρχή του νέου χρόνου. Δυστυχώς, οι, οι προσδοκίες μας δεν επαληθεύθηκαν και όλοι γνωρίζουμε τους λόγους. Το περιεχόμενο των προτάσεων που είχαν τεθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου 2012 και η αναβολή στη συνέχεια των αποφάσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εξάντλησαν τα περιθώρια, ό,τι περιθώρια υπήρχαν για επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας πριν από το τέλος του 2012 η έντονη αντίδραση πολλών συναδέλφων μου υπουργών στην προοπτική σημαντικής μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, την οποία αντίδραση και εμείς ως Κύπρος συμμεριζόμαστε, δεν μας επέτρεψε τελικά να επιτύχουμε τους στόχους μας. Δυστυχώς, επαληθεύθηκαν ταυτόχρονα και οι φόβοι μας ότι η μη επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα σήμαινε και την αναβολή εφαρμογής της νέας ΚΑΠ από 1η 1η 2014. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις για συνέχιση των σημερινών καθεστώτων τουλάχιστον μέχρι την 1η 1η 2015. Παρά τη μη επίτευξη συμφωνίας, η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε σημαντική πρόοδο στα θέματα της ΚΑΠ ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων συναντήσεων και πολιτικών συζητήσεων που είχε οργανώσει και των προτάσεων που είχε υποβάλει σε όλους τους τομείς. Η πρόοδος αυτή καταγράφεται στην έκθεση που ετοιμάστηκε υπό την ευθύνη της Προεδρίας και η οποία σχολιάστηκε πολύ ευμενώς από τις διάφορες αντιπροσωπείες και από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου 2012. Πολλές αντιπροσωπείες επισήμαναν ειδικότερα την αντικειμενικότητα της έκθεσης και την πιστή απόδοση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων που έγιναν. Θα προσπαθήσω τώρα να σκιαγραφίσω σε συντομία την πρόοδο αυτή, αρχίζοντας από την πρόταση κανονισμού για τις άμεσες πληρωμές. Αναφέρω καταρχήν ότι το πρασίνισμα και η εσωτερική σύγκληση των πληρωμών, παρά τη στενή του σχέση με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της εξέτασής τους κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, αναδείχθησαν εν σε κεφαλιώδη θέματα των συζητήσεών μας και τους αποδόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για το πρασίνισμα. Προτείναμε διαδοχικά πέντε προσχέδια αλλαγών και τροποποιήσεων, τα οποία χαιρετίστηκαν από όλες σχεδόν τις αντιπροσωπείες ως βήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Χωρίς να θέτουμε υπό αμφισβήτηση τη βασική αρχή του οικολογικού προσανατολισμού, που είναι το πρασίνισμα όλων των γεωργικών εκτάσεων μιας εκμετάλλευσης, χτίσαμε πάνω στην αρχή της ισοδυναμίας παρέχοντας ευελιξία στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν υπαλλακτικά προς τις τρεις πρακτικές που έχει προτείνει η Επιτροπή διάφορα αγροπεριβαλλοντικά, κλιματικά μέτρα και συστήματα πιστοποίησης με ισοδύναμο περιβαλλοντικό όφελος απλοποιώντας σημαντικά τις αναγκαίες διαδικασίες αντί της εξαίρεσης των ούτω καλούμενων πράσινων εκμεταλλεύσεων εξορισμού που δημιούργησε την εντύπωση ότι επιδιώκουμε πράσινο ξέπλυμα αντιπρασίνισμα εισηγηθήκαμε την εξαίρεση από τη μια ή την άλλη περιβαλλοντική υποχρέωση των εκτάσεων που καλύπτονται από συγκεκριμένες καλλιέργειες και φυτά αναδεικνύοντας έτσι το σημαντικό περιβαλλοντικό και κλιματολογικό ρόλο των μόνιμων βοσκοτόπων, των ψυχανθών, των χορτοδοτικών και υδρόβιων φυτών, των εκτάσεων που περιβάλλονται από δάση και των δεντροδών καλλιεργειών εκτατικού χαρακτήρα. Για τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων εισηγηθήκαμε υπαλλακτικά συστήματα που κατά την άποψή μας διασφαλίζουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα κατά ευέλικτο τρόπο και με χαμηλότερο κόστος. Ασχοληθήκαμε επίσης εντατικά με τη σχέση του πρασινίσματος με τη γραμμή βάσης του δεύτερου πυλώνα και προτείναμε καταρχή λύσεις που ελπίζουμε ότι θα αξιοποιηθούν περαιτέρω. Για το θέμα της εσωτερικής σύγκλησης οργανώσαμε συζητήσεις στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και στο Συμβούλιο και είχαμε εντατικές διμερείς επαφές με όλες τις αντιπροσωπείες. Κατά τη συζήτηση στο Συμβούλιο, πολλοί από τους συναδέλφους μου αναγνώρισαν μεν την ανάγκη για μεταρρύθμιση των ιστορικών πληρωμών και τη σταδιακή σύγκληση, εξέφρασαν όμως επιφυλάξεις για τον χρονικό ορίζοντα και το επίπεδο της επιδιωκόμενης σύγκλησης, ζητώντας γενικά περισσότερη ευελιξία και περισσότερο χρόνο. Τα περισσότερα κράτη-μέλη που σήμερα εφαρμόζουν το ΣΑΠΣ ζήτησαν εξάλλου όπως οι αναεκτάριο πληρωμές διαφοροποιηθούν και στη δική τους περίπτωση ώστε να λαμβάνουν υπόψη και τις άλλες ενισχύσεις που απολάμβαναν οι γεωργοί τους κατά τα τελευταία χρόνια και τούτο έγινε τελικά αποδεκτό από την πλειοψηφία των αντιπροσωπιών. Η Κυπριακή Προεδρία πρότεινε επίσης σημαντικές αλλαγές στα σχέδια για τους νεαρούς και τους μικρούς γεωργούς, οι οποίες έτυχαν πλατιάς υποστήριξης. Για τους νεαρούς γεωργούς προτείναμε μια ενιαία πληρωμή για όλα τα επιλέξιμα εκτάρια της εκμετάλλευσης παρέχοντας ταυτόχρονα στα κράτη-μέλη ευελιξία να καθορίσουν τη δική τους οροφή πέρα από τα όρια που είχε προτείνει η Επιτροπή. Το μόνο σημείο που συνεχίζει να εκκρεμεί για το σχέδιο αυτό είναι ο εθελοντικός ή μη χαρακτήρας του, όπου οι αντιπροσωπείες παρέμειναν διχασμένες. Για τους μικρούς γεωργούς προτείναμε ένα υπαλλακτικό σύστημα που επιτρέπει σε όλους τους γεωργούς που το 2014 θα έπαιρναν κανονικά κάτω από 1.000 ευρώ να ενταχθούν αυτόματα στο σχέδιο, αν το επιθυμούν, και να συνεχίσουν να παίρνουν το ίδιο ποσό μέχρι το 2020. Οι χώρες που προτίθενται να εφαρμόσουν το σχέδιο για τους μικρούς γεωργούς χαιρέτησαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι με το υπαλλακτικό αυτό σύστημα δεν προκύπτει ανάγκη καθορισμού δημοσιονομικής οροφής και μειώνεται η γραφειοκρατία. Η Κυπριακή Προεδρία συμπλήρωσε επίσης τις αλλαγές που έγιναν επί ιδανικής Προεδρίας για την αξιοποίηση των μη δαπανηθέντων ποσών και εισήξε διάφορες βελτιώσεις στον τρόπο κατανομής των δικαιωμάτων πληρωμής παρέχοντας μεταξύ άλλων στα κράτη-μέλη την ευχέρεια να αποκλείουν εκτάσεις που αξιοποιούνται κατά κύριο λόγο από μη γεωργικές δραστηριότητες. Επιτρέψτε μου τώρα να ασχοληθώ σε συντομία με την πρόταση του κανονισμού για την ενιαία κοινή οργάνωση της αγοράς. Στον τομέα αυτό η Κυπριακή Προεδρία διεπίστωσε εξ αρχής ότι οι αντιπροσωπείες ήταν διχασμένες για μια σειρά από σημαντικά θέματα, όπως τα πρότυπα εμπορίας και η επισήμανση του τόπου παραγωγής, η εισαγωγή μηχανισμού για αναθεώρηση των τιμών αναφοράς, η υποχρεωτική αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών των ενώσεών τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων και η επέκταση στα μη μέλη των κανόνων και των εισφορών παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Προεδρίας να επιτύχει συμβιβασμούς, τούτο δεν κατέστη δυνατό με αποτέλεσμα τη διατήρηση του status quo στα περισσότερα από τα θέματα αυτά. Σε μια σειρά από άλλα θέματα, πετύχαμε εν σημαντική πρόοδο. Το πακέτο του γάλακτος ενσωματώθηκε στη βασική πρόταση, βελτιώθηκαν και συμπληρώθηκαν οι πρόνοιες που εισήχθηκαν επί Δανικής Προεδρίας για την ταξινόμηση των σφάγιων και λύθηκαν κάποια προβλήματα στο μελισσοκομικό τομέα. Πολύ θετικό ήταν εξάλλου το γεγονός ότι οι προτάσεις της Προεδρίας <clears throat> για τα έκτακτα μέτρα των άρθρων 154-156 έτυχαν ευρείας υποστήριξης από τις αντιπροσωπείες περιλαμβανομένων και ορισμένων τροποποιήσεων νομικής φύσεως που αφορούσαν την καλύτερη οριοθέτηση των εξουσιών της Επιτροπής να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξης για αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά καθώς και για το περιεχόμενο του όρου Imperative Grounds of Urgency. Τέλος, η πρόταση κανονισμού για την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς προσαρμόστηκε στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών υιοθέτησε τελικά την ερμηνεία της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου για το άρθρο 43.3 TFU e σε ό,τι αφορά τον καθορισμό αποκλειστικά από το Συμβούλιο των τιμών αναφοράς, των τιμών παρέμβασης των ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, του ποσοτικού περιορισμού της βοήθειας για το γάλα στα σχολεία και της ενίσχυσης για το σχέδιο φρούτων στα σχολεία. Η πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών διαφοροποιήθηκε ανάλογα. Είμαι σίγουρος ότι μερικά από τα θέματα αυτά θα επανέλθουν στο προσκήνιο το προσεχές μέλλον όταν θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων. Τώρα, σε σχέση με την πρόταση κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη, θεωρούμε ότι η συζήτηση των εκκρεμούντων θεμάτων, λίγο ή πολύ, ολοκληρώθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας. Ορισμένες αντιπροσωπείες εξακολουθούν εντούτοις να αντιτίθενται ακόμα στην εισαγωγή, έστω και θελοντικά, ταμείου σταθεροποίησης του γεωργικού εισοδήματος κάτω από το δεύτερο πυλώνα, ενώ υπάρχουν άλλες που θεωρούν ότι το κριτήριο απώλειας παραγωγής ή εισοδήματος πέρα του 30% πρέπει να εφαρμόζεται κατά κλάδο παραγωγής και όχι με αναφορά σε ολόκληρη την εκμετάλλευση. Ορισμένες αντιπροσωπείες επιμένουν εξάλλου ότι η συζήτηση για την οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα δεν έχει ολοκληρωθεί παρά την υποστήριξη από την πλειοψηφία των κρατών μελών των προτάσεων της Επιτροπής καθώς και την ευρή αποδοχή της εισήγησης της Προεδρίας για παραχώρηση ενός πρόσθετου έτους για ολοκλήρωση της οριοθέτησης των περιοχών αυτών χωρίς οικονομικές επιπτώσεις. Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε για τα δασικά μέτρα και για τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για βελτίωση της χρήσης του νερού. Η Κυπριακή Προεδρία υπέβαλε μια σειρά από προτάσεις οι οποίες υποστηρίχθηκαν από την πλειοψηφία των κρατών μελών και από την ίδια την Επιτροπή. Σε κρεμότητα παραμένουν μόνο ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που χρειάζεται να αποσαφινιστούν. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μια σύντομη αναφορά στον οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Και στον τομέα αυτό η Κυπριακή Προεδρία έχει επιτύχει βελτιώσεις και σημαντική πρόοδο σε πολυάριθμα άρθρα στοχεύοντας κυρίως στην απλοποίηση και στη μείωση του διοικητικού άχθους. Θα πρέπει εντούτοις να παραδεχτώ ότι η πάγια θέση του Συμβουλίου ότι τα θέματα που σχετίζονται με τους ελέγχους και τις ποινές δεν μπορούν να καθορίζονται με κατεξουσιοδότηση πράξης της Επιτροπής, η συνακόλουθη άρνηση της Επιτροπής να συνεργαστεί για την επεξεργασία λεπτομερών υπαλλακτικών ρυθμίσεων προκάλεσαν σημαντική καθυστέρηση και δυσκολίες τις οποίες η Κυπριακή Προεδρία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μέσα στα δεδομένα χρονικά πλαίσια. Για τον λόγο αυτό, τα περισσότερα άρθρα που σχετίζονται με τις ποινές εντός και εκτός του συστήματος Άγιαξ παρέμειναν σε κρεμότητα μαζί με ορισμένες άλλες πρόνοιες που αφορούν παραδείγματο χάρη τη δημοσίευση των δικαιούχων, το σύστημα ΕΛΠΙΣ σε συνάρτηση με τον οικολογικό προσανατολισμό και προφανώς όλα τα θέματα που σχετίζονται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα να αναφερθώ στα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας και για την υπομονή σας να με ακούσετε. Είμαι τώρα έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας παρακαλώ όμως να περιοριστείτε σε ερωτήσεις που αφορούν την Κυπριακή Προεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Bene, molte grazie Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λετράρη για την ομιλία του και μας απευθύνησε τα σημαντικά βήματα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Και τώρα, όσοι ήθιστε, να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση. Ο κύριος Δες. Παρακαλώ, Άλβερτ. Ευχαριστώ, Παόλο. Κύριε Υπουργέ, ε, Υπουργέ Λετράρη, ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε πάλι στην Επιτροπή μας προσωπικά και εξ ονόματος της ομάδας μου θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά εσάς και όλους τους συνεργάτες σας. Εγώ είμαι πολλά, πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο, έχω δει πολλές προεδρίες και η Κυπριακή συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων των προεδριών που συνεργάστηκε πολύ καλά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρατε πάρα πολλά μέτρα, δεν θα υπησέλθω σε όλα αυτά βέβαια, αλλά μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ένα εξάμεινο περνάει γρήγορα, δώσατε θετική όθηση σε πολλά θέματα και για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος δεν είναι τόσο απλό να προωθήσει όλα αυτά τα μέτρα. Πρέπει λοιπόν να εκφράσω το σεβασμό μου, μεγάλο σεβασμό σχετικά με την ε, Προεδρία σας και την φιλοδοξία που είχατε για την Προεδρία. Μία παράκληση. Εσείς βέβαια θα συνεχίσετε να είστε στο Συμβούλιο. Η παράκλησή μου είναι να προσέξετε πολύ ούτω ώστε να έχουμε γεωργική μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα σε περιοχές ισχνών προϋπολογισμών, ε, που θα βρουν σύμφωνους τους ε, αγρότες στην Ευρώπη. Μέτρα που θα ε, εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, διότι εμείς ε, πρέπει να προσέξουμε πολύ το θέμα της βιωσιμότητας στην Ευρώπη. Υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν, αλλά γενικά πρέπει να είναι λειτουργική και ανταγωνιστική η γεωργία που πρέπει να έχουμε υπόψη μας μια γεωργία που θα τροφοδοτεί όπως πρέπει τα 500 εκατομμύρια κατοίκων μας. Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους πρέπει να δώσουμε στη γεωργία τη δυνατότητα να λειτουργεί όσο γίνεται λιγότερο γραφειοκρατικά, να βοηθηθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι εκμεταλλεύσεις και ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να κάνουν τη δουλειά τους και όχι να κάθονται να συμπληρώνουν έντυπα. Εσείς εργαστήκατε προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω επίσης να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για τις περαιτέρω εργασίες σας. Μάλιστα, ευχαριστώ Άλμπερτ. Ο κύριος Καπλασάντος, παρακαλώ Λουίς. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον ομιλητή. Αγαπητέ κύριε Λετράρη, τους, ε, αυτοί οι τελευταίοι 6 μήνες μας έδειξαν ότι οι καλές προεδρίες δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωγραφική ή με τη δημογραφική διάσταση των κρατών μελών. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τη γενική δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας και θέλω να ευχαριστήσω και σας προσωπικά αλλά και την τεχνική σας ομάδα που βρίσκεται μόνιμα στις Βρυξέλλες είτε τους ανθρώπους από το Υπουργείο σας για το πώς υλοποιήθηκε η εργασία σας αυτούς τους έξι μήνες και για το πώς μπορέσατε να συνεργαστείτε μαζί μας. Η μόνιμη αντιπροσωπεία σας πραγματικά ήταν πολύ συνεργάσιμη στην παροχή επίσημων και άτυπων πληροφοριών και ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμη συνεργασία αυτή την περίοδο που έπρεπε να οικοδομήσουμε και εμείς τη δική μας πρόταση και έπρεπε να εγγυηθούμε ότι οι προτάσεις του Κοινοβουλίου δεν θα απομακρύνονταν σημαντικά από την κατεύθυνση διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου. Εγώ νομίζω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα μας ε, δείχνει ότι οι επαφές αυτές ήταν πάρα πολύ καλές και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το δικό μας θεσμό, για το δικό μας όργανο ο τρόπος ε, που σχετίστηκε η Προεδρία μαζί μας. Και επίση, ε, φυσικά και εσεί, κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε για τη μόνιμη διαθεσιμότητά σα, ε, για τι φορέ που παρευρεθήκατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείξατε ότι σέβεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ και η πολιτική μου ομάδα το εκτιμήσαμε αυτό ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όλοι εμεί που καθημερινά παρακολουθούμε και ζήσαμε όλες ε, αυτές τις μακρές ημέρες εργασίας ε, γιατί εγώ ξέρετε και κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας έζησα αυτά τα πράγματα και ξέρω ότι 31η Δεκεμβρίου είναι μια ευτυχισμένη μέρα πάντοτε για όποιον τελειώνει την Προεδρία και θα ήθελα να σας πω ότι και για το μέλλον θα ήθελα να συνεχίσουμε την επικοδομική συνεργασία, να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιο συμβιβασμό με το Συμβούλιο, γιατί θα είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο για το εξάμεινο που ξεκινά τώρα. Έχουμε ένα δύσκολο στάδιο ενωπιών μας ε, και στο παρελθόν ίσχυε, αλλά και στο μέλλον θα έχουμε ένα δύσκολο στάδιο. Έτσι λοιπόν πάντοτε είναι απαραίτητη μια θετική συνεργασία. Γι' αυτό και πάλι ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ε, σας μεταδώσω και τις προσωπικές μου ευχαριστίες αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Πρόεδρος, ευχαριστώ ο Λουίς, ο κύριος Λάιον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό κύριο λετράρη και την ομάδα του, των συνεργατών του. Ένα θερμό ευχαριστώ από την πολιτική μου ομάδα για το εξαιρετικό έργο και την αφοσίωση που έδειξε αλλά και την ε, επικοινωνία του μαζί μας κατά το εξάμεινο της Προεδρίας. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, υπήρχαν κάποιες ανησυχίε αρχικά σε σχέση με τη μικρή χώρα Κύπρο που αναλάμβανε τόσο μεγάλες ευθύνες αλλά αντιμετώπισαν εξαιρετικά όλες τις προκλήσεις και προώθησαν τα θέματα ε, με πολύ μεγάλη επιτυχία και σίγουρα μας άφησε πολύ ικανοποιημένους η αλληλεπίδραση και η επαφή που είχατε με την Επιτροπή μας. Όλα αυτά ήταν ευπρόσδεκτα. Πάντοτε το Κοινοβούλιο χαίρεται όταν το Συμβούλιο αναγνωρίζει τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε, επειδή είχαμε ψηφοφορίες για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ότι ενδιέφερε πολύ η εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και εκεί το κοινοβούλιο υπήρχε ο φόβος ότι θα επιβράδυνε τις ε, διαδικασίες και αυτό ήταν μια προβληματική δύσκολη. Ενώ εμείς ε, προχωρήσαμε γρήγορα, ενώ φαίνεται να βραδιπορεί το Συμβούλιο. Κολυσιεργούν θα έλεγε κανείς και λέγουν μερικοί. Έτσι λοιπόν δείξαμε ότι είμαστε καλός εταίρος, και είμαστε και πρόθυμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Νομίζω ότι ε, τα παραδοτέα τα είδατε. Είχαμε και καλές συμβιβαστικές ε, λύσεις να προτείνουμε για το Συμβούλιο. Θέλω λοιπόν τέλος να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς εσάς και τους συνεργάτες σας για το έργο σας και για τις επαφές και τη συνεργασία με την Επιτροπή και ελπίζω ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα έχει εξίσου καλή επιτυχία και θα πείσει και το Συμβούλιο να κινηθεί ταχύτερα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Τζόρτζ. Μάρτιν Χόσλιν, παρακαλώ, εξ ονόματος των Πρασίνων. Κύριε Υπουργέ, προσθέτω και εγώ τις δικές μου ευχαριστίες εκείνες των συναδέλφων για την επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή και για το έργο σας. Στην αρχή ε, υπήρχε ε, μια μικρή υποτίμηση όπως ε, υπάρχει και για πολλές άλλες μικρές χώρες, ενώ τώρα ε, θεωρούμε ότι πολλοί άλλοι θα έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας ε, ό,τι αφορά την ε, φιλοευρωπαϊκή στάση. Αυτό είναι βέβαια ένα άλλο θέμα. Κυρίως προσπαθήσατε, πιστεύω, να ξεκαθαρίσετε το θέμα των δημοσιονομικών προοπτικών. Η συνάντηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είχε στεφθεί από ε, επιτυχία, αλλά ε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ε, και το Φεβρουάριο θα γίνει συζήτηση για το θέμα αυτό. Βεβαίως ε, τώρα υπάρχουν εκκρεμότητες μέχρι τη λήψη των δημοσιονομικών αποφάσεων και επειδή υπάρχουν προτάσεις περικοπών και το βλέπετε συμμετέχετε στο Συμβούλιο Υπουργών, αυτό το θέμα των περικοπών το βλέπουμε με μεγάλη επιφυλακτικότητα. Ε, μπορεί ο πρώτος πυλώνας να παραμείνει 100% και να γίνουν μεγάλες περικοπές στο δεύτερο πυλώνα. Αυτό στο μέλλον πρέπει να το αποφύγουμε διότι θα σήμαινε ότι αποστέλουμε λάθος μήνυμα για την κοινή αγροτική πολιτική, ιδιαίτερα στο δεύτερο πυλώνα. Ε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή με τις περικοπές. Εμείς από τη δική μας την πλευρά πρέπει εδώ να εστιάσουμε ε, με μεγάλη προσοχή. Τώρα έχει γίνει ένα βήμα μπροστά, ως ε, ομάδα των πρασίνων ξέρετε βέβαια ότι διαφοροποιούμεθα ε, από πολλούς. Το πρασίνισμα ε, θεωρούμε ότι δεν επιβαρύνει την πολιτική γεωργία στο μέλλον αλλά αποτελεί μια αιτιολόγηση των πληρωμών και στο μέλλον και ελπίζω και η πλειοψηφία στο Συμβούλιο να δει με παρόμοιο τρόπο το θέμα και να μην το θεωρήσει ένα θέμα καθαρά διακοσμητικό. Ε, δεν μπορεί να ε, περιοριζόμεθα στον περιορισμό της ε, γραφειοκρατίας ε, όταν μιλάμε για αγροτική πολιτική, αλλά θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο αποτελεσματικό. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το χρονοδιάγραμμα του έτους αυτού. Εσείς καταβάλατε προσπάθειες ούτω ώστε να μείνουν όλα μέσα στο χρονοδιάγραμμα, στη μεταρρύθμιση. Φαντάζομαι ότι κάποιες καθυστερήσεις θα υπάρχουν, αλλά ελπίζουμε ότι ε, με την έγκαιρη τοποθέτηση του Κοινοβουλίου μπορούμε να προχωρήσουμε στον τριμερή διάλογο και τότε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν από κοινού να φροντίσουν για μια συμφωνία, την επίτευξη συμφωνίας, γιατί ε, σαφώς οι γεωργοί περιμένουν να υπάρξει κάποια σαφήνεια σχετικά με το μέλλον της ε, γεωργικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, πρέπει να καταδείξουμε ε, ε, κατευθύνσεις γρήγορα και στην περαιτέρω διαδικασία ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες διορθώσεις, αλλά ο βασικός προσανατολισμός για την πολιτική γεωργίας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος για το επόμενο εξάμεινο. Ε, νομίζω ότι εδώ θα προχωρήσουμε καλά. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ Μάρτιν. Τζιμ, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ τις ευχαριστίες μου για το, τη σκληρή δουλειά και τις προσπάθειες που καταβάλατε επί της Προεδρίας σας. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά και όλοι αναφέρονται στο γεγονός ότι είστε μικρή χώρα, αλλά μην νομίζετε, πολλές φορές και οι μεγάλοι δεν τα καταφέρνουν καλύτερα. Καμιά φορά τα πάνε και χειρότερα από τους μικρούς. Οπότε συγκρατήστε ότι Κάνατε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό που με ανησυχεί και αναφέρθηκε αυτό, ε, ο Υπουργό δεν θα είναι προεδρεύων, αλλά θα συνεχίσει να είναι στο Συμβούλιο με τους άλλους Υπουργούς Γεωργίας. Και καθώς προχωρούμε προς την ε, ε μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και εμείς μάλιστα την τελευταία μια μισή ημέρα προσπαθήσαμε να ε, τη δική μας τη θέση Πιστεύετε ότι το Συμβούλιο μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του ή θα συνεχίσει να κολλησιεργεί. Θα λάβουν τις αποφάσεις που πρέπει, θα συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο όπως προβλέπει τώρα η συνθήκη της Λισαβόνας ή θα θεωρούν ότι εκείνη είναι η ε, πρώτη τάξη που έχουν βαρύνοντα ρόλο, ε, λόγο. Ε, στην προηγούμενη μεταρρυθμιστική διαδικασία η, ε, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο, αλλά χρειάζεται ε, να παίρνουν το Κοινοβούλιο που τώρα έχει πιο σοβαρό ρόλο πιο σοβαρά. Πιστεύετε ότι θα γίνουν αυτά λέω, σας ρωτώ γιατί δεν θα είστε πια ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, αλλά θα είστε ε, παρόν. Επίσης, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Πριν από λίγα χρόνια, ακούγαμε για την επισητιστική ασφάλεια. Πολλής λόγος γινόταν για αυτό το θέμα. Τώρα δεν το ακούμε πάρα πολύ. Και αναρωτιέμαι, ε, είναι όλα εντάξει εκεί ή μήπως λείπει κάποια πληροφορία, γιατί δεν νομίζω ότι κάναμε ότι ήταν δυνατόν για την επισητιστική ασφάλεια στο μέλλον. Μήπως λοιπόν ε, έχουμε εδώ κάποιο έλλειμμα, μήπως θα εξαρτηθούμε περισσότερο στο μέλλον από εισαγωγές. Πολλοί ανησυχούν ότι τα τρόφιμα και η ε, μεταποίηση ε, στηρίζονται σε πολύ υψηλά πρότυπα, ενώ τα εισαγόμενα πολλές φορές δεν πληρούν τα υψηλά αυτά πρότυπα. Γίνεται ότι είναι δυνατόν ούτω ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της, ε, του εφοδιασμού. Ευχαριστώ. κύριο Άγγλουν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρα Και πάλι καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. Εγώ ε. παρακολούθησα αυτές τις συζητήσεις εδώ τα τελευταία δύο-τρία χρόνια για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. διηρκασαν τεσσερις τέσσερις-πέντε προεδρίες και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς τα πραγματικά γεγονότα ουσιαστικά επισκέψαν τη συζήτηση εδώ. Όταν πρώτα εδώ, άκουγα συνέχεια για την κλιματική αλλαγή και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί μας έλεγαν ε, ότι θα έχουμε πιο ζεστά καλοκαίρια και πιο γρουσιμόνες και κάτι πρέπει να κάνουν οι γεωργοί γι' αυτό. Και μας είπαν ότι θα έπρεπε να βγάλουμε γη από την παραγωγή και θα έπρεπε να κάνουμε και πρασίνισμα. Και αυτό που συνέβη είναι ότι είναι πιο ψηλό ψύχρη χειμωνέ, δείτε και έξω το παράθυρο και είχαμε πραγματικά πολύ υγρά καλοκαίρια. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ε, έγινε δηλώς το αντίθετο. Και τι, τι άλλο έγινε. Και ε, σε σχέση με το 2009 είχαμε αποθέματα σιτηρών σε όλο τον κόσμο, ενώ τώρα έχουμε λήψεις. Και για τρία χρόνια μίλησαμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να αφαιρέσουμε υγεία από την παραγωγή για να ε, δούμε ότι τώρα θα πρέπει να παράγουμε πολύ περισσότερα γιατί δεν έχουμε αρκετό απόθεμα σιτήρων. Εγώ θεωρώ ότι είναι παράδοξο αυτό και χθε ε, είχαμε εδώ μια παραθώνια ψηφοφορία εδώ στην αίθουσα και ε, με ενδιαφέρε που είδα ότι ένας Γερμανός βουλευτής ε, κατέθεσε μία τροπολογία που τα πέταξε όλα, τα κατήργησε όλα και ε, βλέπετε λοιπόν πόση δυσαρέσκεια υπάρχει σε αυτή την επιτροπή. Όμως προσωπικά μου προσφέρατε μία επίσκεψη στην Κύπρο, δεν ε, τα κατάφερα αλλά εκτιμώ την προσφορά και αναρωτιέμαι τι σοδιά είχατε στην Κύπρο πέρσι και τι σοδιά θα περιμένετε να έχετε φέτος το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιξ, παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν, εκ μέρους της ομάδας μου, αλλά και προσωπικά, και εκ μέρους των πολιτών που εκπροσωπώ, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου και να συμφωνήσω με τους προλύσαντες συναδέλφους για τη θετική τους αξιολόγηση. Θα ήθελα όμως να τονίσω κάτι ακόμη. Πιστεύω ότι δεν είναι πολύ καλό να χρησιμοποιούμε όρους όπως μεγάλη χώρα, μικρή χώρα. Όταν ε, ψήφισαν οι πολίτες μας για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αναφερθήκαμε στο μέγεθος των κρατών μελών. Ε, ξέραμε ότι όλα τα κράτη-μέλη είναι ίσα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, υποσυνείδητα υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των μικρών και των μεγάλων χωρών και φαίνεται σαν να αισθάνονται μικρές χώρες ότι ε, πρέπει να ακολουθούν τις μεγάλες. Ε, όμως, κύριε Υπουργέ, προερχόμενος από αυτό το μικρό κράτος μέλος ε, δείξατε παρόλα αυτά ισχύει και δείξατε ότι μια μικρή χώρα μπορεί να δράσει με τον ίδιο τρόπο όπως και τα μεγάλα κράτη-μέλη μας δείξατε ότι μπορείτε να πετείτε σεβασμό από όλους τους υπολείπους και όλοι σας είπαν ευχαριστώ για το έργο σας. Επίσης, ε, θέλω να πω ότι η στάση σας ήταν πάρα πολύ ανοιχτή και το ίδιο ισχύει για τους συναδέλφους σας ε, από την Κύπρο και αυτό το εκτιμώ. Πάντοτε ήσασταν έτοιμοι να μας ακούσετε, να συνομιλήσετε μαζί μας και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Βεβαίως, ε, όταν ξεκίνησε η Προεδρία σας, όλο θέμα της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής ε, είχε αρχίσει να φτάνει στο τελικό του στάδιο. Επομένως ήταν πάρα πολύ δύσκολο το δικό σας έργο και είχε και μεγάλες ευθύνες. Εγώ πιστεύω ότι κάνατε πολύ καλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά προφήσατε την ε, μεταρρύθμιση και φυσικά αυτό μπορεί να αποτελέσει μια βάση για τη δουλειά των επόμενων Προεδριών. Και βέβαια πάντοτε θα γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ και μεγάλων χωρών ε, και όσων θέλουν να πετύχουν, το τάδε το δίνα. Όμως ε, εμείς σας ευχαριστούμε που προωθήσατε την όλη διαδικασία και εκ μέρους ε, των πολιτών θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι οι άμεσες πληρωμές θα είναι δύο φορές μεγαλύτερες από παλιά. Βέβαια έχουμε μόνο τα δύο τρίτα του μεσουόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γεωργοί πάντοτε με ρωτούν ε, πότε πρέ, πόσο καιρό πρέπει να περιμένουμε για να υπάρχει απολύτη Από ό,τι καταλαβαίνω όμως δεν εξαρτάται αυτό μόνο από εσά, αλλά εμείς αισθανόμαστε τα όσα έχουν επιτευχθεί στην παραγωγή του τομέα της ζάχαρης, παραδείγματος χάρη και στη διατήρηση των ποσοστώσεων στη ζάχαρη. φαίνεται σαν να υπάρχει προστατευτισμός από τους μεγάλους παραγωγούς ε, ζάχαρης. Όμως είναι ικανοποιημένοι με την ποσόστοση που τους δόθηκε. Εγώ πιστεύω ότι την εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση τους καιρού που η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε εισαγωγή ζάχαρη και ενώ υπάρχει έλλειψη ζάχαρη στον κόσμο και το ίδιο και για το γάλα, φαίνεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είμαστε σε θέση να παράξουν οι γεωργοί μας ε, τα προϊόντα που χρειάζονται να τα αποθηκεύσουμε και να τα προσφέρουμε κατόπιν όταν υπάρχει ανάγκη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάνω από 800 800 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίω που ζουν ε, σε συνθήκε φτώχεια. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πάντως εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσουν και οι υπόλοιποι να εργάζονται με το ίδιο πνεύμα που δείξατε εσεί. θα πετύχουμε πολλά. Σα. ευχαριστώ για τη συνεργασία. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε τον γύρο παρεμβάσεων. Όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων πήραν το λόγο. Εγώ και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λετράρη για το έργο που υλοποίησε ως ε, πρόεδρος του Συμβουλίου Γεωργίας και θα του δώσω το λόγο για κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές. Είναι αλήθεια ότι η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, πρέπει να το ομολογήσουμε, με πολύ περιορισμένους πόρους και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε λεφτά. Ήταν η πρώτη φορά που αναλαμβάναμε την Προεδρία του Συμβουλίου και νιώθαμε μεγάλη την ευθύνη. Γι' αυτό δουλέψαμε με ενθουσιασμό και με επαγγελματισμό για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που τα οποία αναφερθήκατε για την Κυπριακή Προεδρία πραγματικά με, με συγκίνησε διότι τόσο καλά λόγια κάποιος ακούει μόνο στον επικίδιο του όταν έχει πεθάνει και μιλάνε άλλοι γι' αυτόν. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αναφέρθηκε ο κύριος Δες ότι υπάρχει ανάγκη η η μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής να βρει σύμφωνο στους αγρότες μας και ήταν πάντα που το τόνιζα αυτό όταν άκουγα για μερικές προτάσεις που ήταν έτσι μη ρεαλιστικές, εξωπραγματικές ότι πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα τον γεωργό, τον αγρότη αυτό τον οποίο απευθύνεται η ΚΑΠ. Σίγουρα το περιβάλλον έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει αλλά ο αγρότης, ο γεωργός, είναι η σημαντικότερη συνιστόσα της εξίσωσης. Και αν θέλουμε να έχουμε μια λειτουργική, ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία, θα πρέπει η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να κινηθεί σε αυτά τα πλαίσια και προπάντων, προπάντων απ' όλα, χωρίς γραφειοκρατία. Πραγματικά το Υπουργείο, το δικό μου στην Κύπρο, και ειδικά τα τμήματα που ασχολούνται με την ΚΑΠ αναλώνουν τον χρόνο τους γεμίζοντας έντυπα και φόρμες και ετοιμάζοντας εκθέσεις με ένα τρομερό διοικητικό κόστος. Οπότε αν επιβάλλεται όπου μπορούμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Ε, σίγουρα ήταν χρήσιμες οι επαφές που είχαμε μεταξύ μας για να γνωρίσετε και εσείς την θέση περίπου που πάει να κινηθεί το Συμβούλιο, αλλά και εμάς για να προσαρμόσουμε τις δικές μας θέσεις σαν Συμβούλιο ανάλογα με το που κινείται το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν έχει έννοια μεγάλη εάν κινούμαστε σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρεθούν συγκλήσεις. Από την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκα κοντά σας ανάφερα ότι εμείς σεβόμαστε το Ευρωκοινοβούλιο και τον, ε, το ρόλο του, τον αναβαθμισμένο ρόλο του σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε μπροστά μας τώρα ένα αρκετά δύσκολο εξάμεινο. Έχουμε όμως κάτι πιο ξεκάθαρο, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένω ότι η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου θα υιοθετήσει τις δικές σας αποφάσεις άρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους συμβιβασμού. Ε, επειδή αναφερθήκατε σε πιθανή κόλληση εργία του Συμβουλίου και για το κατά πόσον το Συμβούλιο δέχεται την, το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου για τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να πω ότι η ευθύνη οποιασδήποτε Προεδρίας και της Κυπριακής Προεδρίας ήταν να εκφράζει με ένα πιστό και αντικειμενικό τρόπο τις θέσεις της πλειοψηφίας του, των κρατομελών και αυτό ακριβώς ε, κάναμε. Είναι γεγονός ότι το Συμβούλιο αισθάνεται έντονα σε μερικά θέματα και είναι γνωστό το γεγονός αυτό. Είναι θέμα πραγματικά διαπραγματεύσεων και πιστεύω ότι όλες οι πλευρές θα προσέλθουν με καλή θέληση και με ανοιχτό μυαλό την ευθύνη τώρα για τους περαιτέρου χειροσμούς την έχει η Ορλανδική Προεδρία και της εύχομαι κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι ο συνάδελφος μου, ο Ιρλανδός Υπουργό θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά. Ε, ναι, μας στενοχώρησε ιδιαίτερα ότι δεν επήλθε κάποια συμφωνία στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ήταν αλήθεια ότι στη φάση εκείνη η Υπουργοί Γεωργίας ήταν ε, έτσι πολύ αναστατωμένη και πολύ δυσαρεστημένοι με την εξέλιξη αυτή σε σημείο μάλιστα που να μην θέλουν καν να συνεχίσουμε και να κάνουμε περαιτέρω πρόοδο σε κάποια θέματα που είμαστε κοντά. Ε, να διαβεβαιώσω τον κύριο Χόσλινγκ ότι το πρασίνισμα είναι πολύ σοβαρό θέμα, σε καμιά περίπτωση δεν είναι διακοσμητικό και θα έλεγα χωρίς εξαίρεση όλα τα κράτη-μέλη και όλες οι αντιπροσωπείες το παίρνουν στα σοβαρά και το επιθυμούν αλλά όπως και να το κάνουμε εάν ζητούμε από τους γεωργούς να εφαρμόσουν κάποια πρόσθετα μέτρα θα πρέπει και ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ να είναι ανάλογος και υγιής προϋπολογισμός. Ε, αναφερθήκατε στην επιστημιστική ασφάλεια και διαρωτηθεί ε, και ο κύριος Νίκολσον εάν είναι όλα εντάξει. Όχι, είναι φανερό ότι έχουμε λύματα, ε, εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό και θα εξαρτόμαστε και στο μέλλον από εισαγωγές, ε, αλλά ο σκοπός της ΚΑΠ είναι ακριβώς να επιλύσει και αυτό το πρόβλημα, κάνοντας τη γεωργία μας ανταγωνιστική μην ξεχνάτε ότι πολλές εισαγωγές γίνονται ακριβώς γιατί τα ευρωπαϊκά μας προϊόντα που είναι καλύτερα και με πιο αυστηρά πρότυπα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά όσο τα προϊόντα άλλων κρατών, τρί, τρίτων χωρών εννοώ. Ε, ο κύριος Άχνιο αναφέρθηκε στις κλιματικές αλλαγές. Είναι αλήθεια ότι μας προβλημάτισε το γεγονός αυτό. Ε, στο άτυπο Συμβούλιο που διοργανώσαμε στην ε, Λευκοσία το, το Σεπτέμβριο ήταν το κύριο μας ε, θέμα κλιματικές αλλαγές και επιστημιστική ασφάλεια, χρήση των πόρων, ειδικά των υδάτινων πόρων ε, και είναι κάτι που μας προβληματίζει πάρα πολύ. Αλλά κλιματικές αλλαγές δεν σημαίνει όπως το έχετε πει πιο υγρά καλοκαίρια και περισσότερα χιόνια, κλιματικές αλλαγές για μας που είμαστε στον Νότο σημαίνει ξηρασία, ανοβρία και αύξηση της θερμοκρασίας. Επειδή ερωτηθήκατε για τη σοδιά μας φέτος στην Κύπρο, είχαμε μια πολύ καλή χρονιά όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Ευτυχώς τα φράγματα μας στο νησί είναι σχεδόν ε, πλήρη, είναι γεμάτα, υπερχιλίζουν τα περισσότερα αλλά αυτός δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι τα φράγματα μας είναι άδεια λόγω των κλιματικών αλλαγών και οι σοδιές μας δεν είναι πάντα τόσο καλές. Όσον αφορά την επίσκεψη που σας προσκάλεσαν να έρθετε στην Κύπρο, ισχύει και θα ισχύει πάντοτε. Ε, κύριε Πρόεδρε, εν ολίγης αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία ναι, για όλους τους ευρωβουλευτές, ειδικά για σας κύριε Πρόεδρε που είστε, ήσασταν πάντα διαθέσιμος για συναντήσεις. Είμαι σίγουρος ότι και στο μέλλον θα υπάρχει η ίδια και καλύτερη συνεργασία με την Ιρλανδική Προεδρία για το καλό της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ. Bene, colleghi, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συνεδρίασή μας την επόμενη εβδομάδα στις 31, 9 το πρωί. Θα συναντηθούμε για να ανταλλάξουμε απόψεις με το νέο ε, πρόεδρο του Συμβουλίου, τον Ιρλανδό Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Κόνη.